Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Ε, πρέπει να περιμένω μία επιβεβαίωση από το Προεδρείο ότι ε, ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε όντως είχε εγκριθεί από το Προεδρείο. Αυτό όντως έλαβε χώρα και μου διαβιβάστηκαν και τα σχετικά έγγραφα. Ήσασταν παρόν, έτσι δεν είναι. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, μπορούμε να εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη. Στα παραρτήματα 1 και 2 έχετε το περιεχόμενο συμβασμού αυτού που θα τον ψηφίσουμε το σε λίγο. Λοιπόν, οι αποφάσεις των συντονιστών της συνεδρίασης ε, της 21ης Μαρτίου βρίσκονται στο φάκελό σας. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση θεωρώ ότι εγκρίνονται. Προτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για το σχέδιο προπολογισμού για το Κοινοβούλιο για το έτος 2019. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Αιντέρ Καρθιαμπάλ Ρουμπιάλ για την περίπτωση της Caterpillar και την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα γρήγορα γιατί έχουμε μετά ψηφοφορίες οι οποίες χρειάζονται αρκετό χρόνο. Έχουμε ένα νέο αίτημα όπως είπατε και εσείς για το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Υπέβαλαν το αίτημα αυτό οι αρχές του Βελγίου λόγω των απολύσεων στο εργοστάσιο της Caterpillar. Το 2015 για την είδα για εταιρεία είχαμε αίτημα 1.300 απολύσεις με το ποσό με το οποίο αποζημιώθηκαν και φέτος έχουμε ένα πολύ υψηλότερο αίτημα αποζημίωσης ε, για 2.287 απολυμμένους ε, που θα μας φέρει σε ένα ποσό 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Ε, έχουν ε, μειωθεί αυτές τις εργασίες γιατί μειώθηκαν οι εξαγωγές, γιατί αυξήθηκε το κόστος παραγωγής, γιατί έχουμε την ε, εντατική, τον εντατικό ανταγωνισμό από τις επιχειρήσεις στην Κίνα. Παρόλα αυτά πρέπει να πω πως αυτή η εταιρεία παρόλο που έκανε αυτές τις απολύσεις ήταν μια επιχείρηση με κέρδη και μάλλον επρόκειται για μια επιχειρηματική απόφαση ε, στρατηγικής που να κλείσει αυτό το εργοστάσιο. Να σας πω πως ε, ε, τέτοιου είδους απολύσεις μας δημιουργούν απέχθεια, αλλά ο στόχος μας είναι μέσω των κονδυλίων του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση να διευκολύνουμε τους απολυμμένους εργαζόμενους έτσι ώστε να ξαναμπούν το συντομότερο δυνατό στην αγορά ε, εργασίας. Δηλαδή να τους βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό, να περάσουν από εκπαίδευση και να συνεργαστούμε με τοπικές αρχές. Και επίσης κάποιες επιδοτήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στήριξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ανθρώπων αυτών, για την εκπαίδευση και για την δυνατότητα απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Νομίζω πως το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αυτούς τους απολυμμένους εργαζόμενους, αλλά και για άλλα 300 νεαρά άτομα που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή ούτε σε συνθήκες εκπαίδευσης, ούτε σε συνθήκες εργασίας. Άρα λοιπόν στην έκθεσή μου αυτά περιγράφω και ελπίζω να ακούσω τώρα και τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεπρέ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την συνάδελφο για την ποιότητα αυτής της έκθεσης η οποία μας έχει καταθέσει και που θα σας ε, καλέσω να στηρίξουμε. Απλώς θα ήθελα να μιλήσω για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Η Caterpillar ήταν ένα εργοστάσιο πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή του Σαρλερουά, η οποία είναι μια περιοχή η οποία έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλη ε, βιομηχανική ε, αναδόμηση, γιατί χάσανε τη χαλιβουργία, χάσανε την επεξεργασία ε, μεταλλικών στοιχείων, έχουν 52% επίπεδα ανεργίας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και βέβαια στην ε, επαρχία του ΕΝΟ το ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο στην Ευρώπη παρόλο που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης. Οπότε αυτή η εταιρεία είχε περάσει με τα ε, αναδιάρθρωση το 2013 και το 2014 και το, μέχρι το 2015 η Caterpillar δεν έκανε καμία επένδυση και το 2016 με μια απλή ανακοίνωση η πολυεθνική από τη ΣΥΠΑ ανακοίνωσε απλώς πως κλείνει το εργαστήριο εργοστάσιο χωρίς να διαβουλευτεί το θέμα αυτό με τις βελεϊκές αρχές και φέρει την καταστροφή στην περιοχή. Δεδομένων λοιπόν των περιφερειακών ε, προβλημάτων, οι περιφερειακές αρχές προσπάθησαν να ξεκινήσουν κάποια προγράμματα ε, επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για να βρει ε, δουλειά. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε κάποια από τα αποτελέσματα του τι φέρνει η παγκοσμιοποίηση και το τι συμβαίνει με τέτοιου είδους αναδιάρθρωση που φέρνει το βαρύ τίμημα της ανεργίας με πολλά προσωπικά προβλήματα που για τους εργαζόμενους είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Νομίζω το δεύτερο κύμα αιτήματο ε, ε, ε, δεύτερο κύμα απολύσεων από την Caterpillar, αν δεν κάνω λάθος. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα σου από τους συναδέλφους. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε δική μας χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά και λογικά. Για παράδειγμα, νομίζω ότι θα πρέπει να προβλεφθούν τα απαραίτητα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, να καταφέρουμε να προτιμάσουμε τους απολυθέντες εργαζομένους για νέα σχέδια επιχειρηματικότητας, να βοηθήσουμε τους νέους να δημιουργήσουν νέες νεοφυείς επιχειρήσεις. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει επίσης να εμπλεκούν και οι ε, εθνικές αρχές ε, του Βελγίου. Οι δημόσιες αρχές και αρχές της Βαλωνίας θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσουν το σχέδιο αυτό. Αυτό θα γίνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν είναι χαμένα χρήματα σε καμία περίπτωση, αλλά θα πρέπει σίγουρα να έχουν ω απότερο στόχο να ενταχθούν εκ νέου οι απολυθέντε εργαζόμενοι τη Caterpillar στην αγορά εργασία. Πολύ ωραία, δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Να σα διευκρινίσω ότι μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, οι τροπολογίε θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 18 Απριλίου 12 το μεσημέρι, δηλαδή την Τετάρτη το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 23 Απριλίου και θα περάσει το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια στις 3 Μαΐου. Πρόκειται για μήνυ Ολομέλεια που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σχέδιο προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση πάντρουμπικα. Σας παρακαλώ πολύ Βάλτε τώρα τις κάρτες σας στις συσκευές ψηφοφορίας για να κάνουμε μια πρώτη δοκιμή. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Πολύ ωραία. Παράρτημα 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράρτημα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι 12, 13, 14 καταπίπτουν διότι εγκρίθηκε από το Προεδρείο το κείμενο και από την ψηφοφορία που είχαμε τώρα, τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 και 22 από κοινού υπέρ. Κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για τις τροπολογίες 21 και 22. Άρτη ψηφοφορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την κάρτα της κυρίας Στομά. Λειτουργεί ή όχι η συσκευή. Λειτουργεί. Πολύ ωραία. Πέρασε. εγκρίνεται 24 υπέρ 13 κατά Ψηφίσαμε στις τροπολογίες 21 και 22. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 23. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 καταπίπτει. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 43 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, διορθώνει ο Πρόεδρος. Η 44 τώρα παρακαλώ, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 47. Πέρασε. Απορρίπτεται 22 με 37. Λοιπόν, 48 υπέρ κατά απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 με μία τροπολογία προφορική υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται βλέπετε 37 με 21. Καταπίπτει 50, η 60 καταπίπτει, 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 καταπίπτει. 52 με τεχνική προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 καταπίπτει 58 καταπίπτει 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 με προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω απερίπτεται το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. 37-19. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για τη συμβιβαστική 3 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19-15. Προφορική τροπολογία του κυρίου Ρούμπιχ για την 25α υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται συν 18 μείον 20. 66 υπέρ. 76 με συγχωρείτε υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Είμαστε στην 76. Έχετε ψηφίσει όλοι. Κάποιος λείπει. Πέρας. Εγκρίνεται. 22-14. 77 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική υπάρχουν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 82 έχει αποσυρθεί περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία της κυρίας Γκουαρδία Ζαμπάλ και των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ πολύ άρχεται η ψηφοφορία όλοι δύο δεν έχουν ψηφίσει πέρας εγκρίνεται 18-16 90 υπέρ αποχές εγκρίνεται. Προφορική του κυρίου Ρούμπιχ. Είναι για την παράγραφο 27α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Πρέπει όμως να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας λείπει. Πέρας. Απορρίπτεται. 15-21. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 είναι προφορική τροπολογία της κυρίας Γκαρδίας Άμπαλ από τους σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά θα το επαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά ε, ξεκινάει η ψηφοφορία Κάποιος από εσάς πάλι δεν έχει ψηφίσει. Πέρας. Εγκρίνεται 21, 15 και 2 εποχές. Περνάμε τώρα στην 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Έχουμε 40 κάρτες και 38 ψήφους. Απορρίπτεται. 24-12. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102. Με προφορική τροπολογία του κυρίου Χάουαρθ από τους σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 105 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Από το ΕΛΚ έχουμε μία παραπάνω. Ποιος είναι. Πέρας. Εγκρίνεται. 23-14. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 108, 109, 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην 111 καταπίπτει και περνάμε στην 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στα εκτιμώντας. Υπάρχει μόνο ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία.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 7 και 8 έχουν τον ίδιο στόχο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 9. Είναι τεχνική που δεν χρειάζεται ψηφοφορία. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και φτάσαμε λοιπόν στην συνολική ψηφοφορία για όλο το κείμενο. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 33 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια, κύριε Ρούμπιχ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για όσους από εσάς είχατε τύψεις γιατί δεν ήρθατε στην συνάντηση των ελέγχων των προπολογισμών να σας πω πως αυτή τη στιγμή συνεδριάζει στο ΒΙΚ 200 η Εν Λόγω Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Θέματα για τα διάφορα δεν βλέπω. Λύεται η συνεδρίαση.